Καλησπέρα συνάδελφοι. Να σας καλωσορίσω στην απογευματινή συνεδρίαση. Λέγομαι Ντίτα Χαράντσοβα. Είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδια για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και επομένω να σας καλωσορίσω θερμά και εγώ από πλευράς μου και είναι τιμή μου που προεδρεύω σήμερα το απόγευμα στη συζήτηση αυτή. Με πολύ χαρά καλωσορίζω εδώ και τον άλλο ε, συμπρόεδρο, τον κύριο Μάρας, ε, πρόεδρο της ε, Επιτροπής Εργασίας, Συνταξιοδότησης και Κοινωνικής Συνοχής του Κροατικού Κοινοβουλίου, που θα συμπροεδρεύσει μετά από την εισαγωγή μου. Όπως γνωρίζετε, Εδώ επικεντρωνόμαστε σε δεξιότητες και θέσεις εργασίας για μια ανάπτυξη που περιλαμβάνει τους πάντες και τι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από την εμπειρία του άλλου. Όπως γνωρίζετε, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις ολοένα ε, μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας ήταν ε, μια ε, πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέκαθεν και είναι και πάρα πολύ σημαντική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην προηγούμενη το Κοινοβούλιο ενέκρινε αρκετές, ε, αρκετά συγγνώμη, σχετικά ψηφίσματα για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας για τον 21ο αιώνα και ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, επιμένοντας για την ανάγκη να αναπτύξουμε ή να αναβαθμίσουμε δεξιότητες διαβίου και να, για θέσεις εργασίας και να τονίσουμε και το ρόλο της εκπαίδευσης και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση. Επίσης, όπως όλοι γνωρίζουμε, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εθνική αρμοδιότητα. Επομένως, είναι ζωτική σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ακούσουν και τις απόψεις των εθνικών μελών των κοινοβουλίων ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές μας θα είναι συμπληρωματικέ στα εθνικά σχέδια δράσης και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε όπου χρειάζεται προκειμένου να προσαρμοστούμε σε αυτόν τον κόσμο που συνέχεια αλλάζει. Με αυτές τις σύντομε παρατηρήσεις λοιπόν θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον συμπρόεδρό μου, στον κύριο Μάρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε Χαραντσόβα, Αγαπητοί συνάδελφοι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελπίζω ότι σήμερα θα έχουμε μια καρποφόρα συζήτηση για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι οι δεξιότητες και οι θέσεις εργασίας για την ανάπτυξη που περιλαμβάνει τους πάντες είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον πρώτο ομιλητή από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, ο Επίτροπος για τις θέσεις εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα για να κάνει κάποιες πρώτες παρεμβάσεις, ο κύριος Νίκολας Σμιτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές. Οι ταξιότητε αποτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο για την ε, βιώσιμη και ευρεία ανάπτυξη σε ό,τι αφορά και την ε, ψηφιακή μετάβαση. Είναι πολύ επίκαιρη η σημερινή συνεδρίαση, γιατί σήμερα το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά από σημαντικές στρατηγικές. Η στρατηγική για την ψηφιακή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια λευκή βίβλο επίσης για την τεχνητή νοημοσύνη και ένα έγγραφο για τα δεδομένα. Είναι σωστή λοιπόν η σημερινή στιγμή να συζητήσουμε το θέμα των δεξιοτήτων. Γιατί σε όλους αυτούς τους πολύ σημαντικούς τομείς οι δεξιότητες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο. Και θα πετύχουμε την ψηφιακή μετάβαση μόνο εφόσον και αν προετοιμάσουμε τον κόσμο για την ψηφιακή αυτή επανάσταση. Άρα, επιλέξατε το σωστό θέμα τη σωστή στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν εργαζόμαστε σε θέματα ψηφιακής μετάβασης. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε στην αρχή της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ατζέντα για τις δεξιότητες και τις ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη αρχή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικά κενά και αναντιστοιχίες σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες και πάνω από 30% των ε, Ευρωπαίων δεν έχουν τη σωστή ψηφιακή τον ψηφιακό αλφαβητισμό και τις δεξιότητες που χρειάζεται. Και πάνω από 90% των θέσεων απασχόλησης πλέον προϋποθέτει μια κάποια ένα κάποιο επίπεδο ψηφιακής δεξιότητας, καθώς και η συμμετοχή γενικά στην ε, κοινωνία τεχνητή νοημοσύνη, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η συμμετοχική δημοκρατία, όλα αυτά προποθέτουν κάποιε βασικέ δεξιότητέ. Και σύμφωνα όμω με την σχετικό δίκτυο για την ψηφιακή οικονομία για το 2017 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, 43% του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει ανεπαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και 17% δεν έχει κανένα επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Και προφανώ οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν να βρεθούν σε θέσεις ανεργίας. Μεταξύ του 2012 και 2016 η απασχολησιμότητα των ανθρώπων αυτών μειώθηκε κατά 10%. Αυτό όμως δεν είναι το βασικό και μόνο πρόβλημα. Τίφεται και θέμα αποτελεσματικής ε, διάδρασης με πολλές υπηρεσίες ε, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες υγείας για παράδειγμα ακόμα και μέχρι και τις αγορές online. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με την οικονομική και την κοινωνική διάσταση και θα πρέπει να επενδύσουμε στις δεξιότητες για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Μεγάλα ζητήματα όπως η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, οι οικονομίες συνδενικού άνθρακα θα προϋποθέτουν δραστηριότητες και δράσεις σε όλες τους ε, τομείς για να υπάρξει προσαρμογή των νέων αυτών δεξιοτήτων που θα χρειαστούν από το εργατικό δυναμικό. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι το εργατικό δυναμικό θα πρέπει να επανακαταρτιστεί τα επόμενα χρόνια. Και αυτό κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι εκείνες που πλήττονται πιο πολύ από την ψηφιακή μετάβαση 79% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δήλωσαν ξεκάθαρα ότι χρειάζονται τουλάχιστον τις ε, θεμελιώδεις βασικές ε, ψηφιακές δεξιότητες και το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την ε, κατάρτιση του προσωπικού τους είναι το οικονομικό κόστος. Η πρόκληση λοιπόν είναι τεράστια. Δεν υπάρχουν πλέον οι δουλειές για μια ζωή. Οι πολίτες κάνουν 10 και παραπάνω αλλαγέ καριέρα. Αλλαγέ, μάλλον θέσεις απασχόληση στην καριέρα τους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην αγορά εργασία. Προκειμένου λοιπόν η κινητικότητα αυτή να καταστεί μια ευκαιρία για όλους, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος έχει και μια αίσθηση ασφάλεια. Ασφάλεια σημαίνει ότι θα του συνοδεύσουμε σε αυτέ τι ε, αλλαγέ. Ένα σημαντικό λοιπόν θέμα είναι οι δεξιότητε. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι ένα εξασφαλισμένο εισόδημα. Και τρίτον, προφανώ θα χρειαστεί και κάποια καθοδήγηση, γιατί είναι εύκολο να λέμε σε κάποιον άλλαξε δουλειά και φρόντισε να αποκτήσεις διαφορετικές δεξιότητες. Αλλά στην ουσία ο κόσμος για να πετύχει χρειάζεται κάποια καθοδήγηση. Για να πετύχουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτό, χρειαζόμαστε νέε πολιτικέ οι οποίε θα βάλουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Τονίζοντα ε, και την κοινωνική και συλλογική ευθύνη όλων των εμπλεκομένων φορέων. Γι' αυτό λοιπόν σκοπεύουμε να ενδυναμώσουμε την ατζέντα για τι δεξιότητε. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πάνω απ' όλα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και κυρίως με τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους θα υιοθετηθεί σχετική ανακοίνωση τέλη Μαρτίου. Η ενημερωμένη λοιπόν ατζέντα για τις δεξιότητες έχει τρεις βασικούς στόχους. Καταρχάς, η ενδυνάμωση των εργαζομένων και των ε, υπαλλήλων για να κάνουν ε, εκ νέου κατάρτισης. Κατά δεύτερον, στρατηγική σχετική από τις επιχειρήσεις ε, για το εργατικό δυναμικό με την οικονομική δέσμευση που συνεπάγεται και κατά τρίτον για να είμαστε επιτυχείς θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια σειρά κρίσιμων δράσεων για να πετύχουμε τις ε, αλλαγές οι οποίες χρειάζονται τόσο πολύ. Όταν μιλάω για αλλαγές μιλώ και για την ατροπία. Θα πρέπει να δείξουμε ότι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εναλλακτικών δεξιοτήτων δεν αποτελεί με υποχρέωση μόνο, αλλά και μια ευκαιρία όσο αλλάζει λοιπόν το περιβάλλον εργασία, όσο αλλάζουν και οι δουλειέ. Η αλλαγή θέση μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για τον κόσμο. Γιατί η νέα αυτή θέση απασχόληση ενδεχομένω να είναι λιγότερο δύσκολη περίπλοκη σε σχέση με την προηγούμενη. Το Μάρτιο λοιπόν θα υποβάλουμε μια πρόταση για τις συστάσεις του Συμβουλίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα εξυγχρονίσει την ευρωπαϊκή πολιτική κάνοντας τη σύνδεση με τις ψηφιακές ε, τεχνολογίες και την ψηφιακή μετάβαση. Επίσης ενίσχυση του Εράσμους και ενίσχυση της διαβίου μάθησης σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση. Και μία κοινή φιλοδοξία που θα πρέπει να έχουμε είναι να αξιοποιήσουμε την επαγγελματική κατάρτιση. Γιατί αυτό θα βελτιώσει και τη δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών δεξιοτήτων. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη λοιπόν διανομή των πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει πραγματικά ανάγκη για διαφορετικές δεξιότητες για όλους. Αλλά να έχουμε υπόψη ότι ο πιο πολύ κόσμος αναπτύσσει έτσι κι αλλιώς νέες δεξιότητες. Αυτές οι εμπειρίες ωστόσο όμως συχνά δεν αναγνωρίζονται και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ενδεχομένως όπως θα έπρεπε. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε προσοχή. Και όλος ο θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στο άτομο για να μην ακυρωθεί η αξία του να δώσουμε προσωπικό, προσωπικές συμβουλές, οικονομικές, ε, οικονομική ενέσχυση για να υπάρξει καλύτερη αναγνώριση των ε, σημαντικών δεξιότητων τους. Και έχουμε τα ευρωπαϊκά λοιπόν ταμεία για να τα υποστηρίξουμε όλα αυτά. Ήδη έχουμε κάποια καλά παραδείγματα. Για να αναπτυχθούν λοιπόν σχετικές πολιτικές σχετικά με τη δεξιότητα και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κάποιες ε, χώρες έχουν μεταρρυθμίσει την επαγγελματική κατάρτιση και το σχετικό σύστημα πιστοποίησης. Άρα, κλείνοντας, να πούμε ότι χρειάζεται αποτελεσματική επένδυση σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει η Ευρώπη να δαπανίσει και να επενδύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να επικεντρωθούν αυτές οι επενδύσεις και να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία για μια αποτελεσματική στρατηγική για τις δεξιότητες. Ελπίζω μέσω της συζήτησης που θα γίνει τα μηνύματα αυτά να ληφθούν υπόψη τα κοινοβούλια σας, γιατί σε τελική ανάλυση στα κράτη-μέλη επαφίεται να δώσουν επιτυχία και πνοή σε αυτή την στρατηγική της δεξιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σμέτε για την παρέμβασή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας ε, στηρίξατε εχθές ε, και σήμερα στις Επιτροπές. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά σας και ευχαριστούμε πολύ για τα εισαγωγικά σας ε, σχόλια. από τη Φινλανδία, η κυρία Κιλόινεν είναι αντιπρόεδρος της αρμόδιας της Επιτροπής Δανειοδοτήσεων του Φινλανδικού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές για την οργάνωση αυτής της συνεδρίασης. Ε, είναι χαρά μου το ότι μπορώ να σας μεταφέρω κάποιες απόψεις από τη Φινλανδία που ελπίζω να χρησιμεύσουν ως σημείο κίνησης για περαιτέρω συζητήσεις. Ε, πραγματικά βρισκόμαστε στο μέσο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, μια επανάσταση που χαρακτηρίζεται από την ψηφιοποίηση, την όλο μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση ε, και πολιτικές οι οποίες ε, συζητιούνται ε, για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να αμβληνθούν οι επιπτώσεις. Η ψηφιοποίηση θα διευκολύνει τη ζωή μας, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης σε όλους τους τομείς της ζωής και στην παιδεία και νομίζω μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τώρα πια ο κόσμος είναι ε, το κουκούλι μας με την έννοια ότι ακόμα και οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους ε, και να διευρύνουν την ε, αγορά τους. Ε, το αρνητικό στοιχείο είναι ότι θα εξαφανιστούν οι παραδοσιακές θέσει απασχόλησης. Πολλοί ε, θα κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους ε, και Τώρα, ποιο θα ωφεληθεί από τις αλλαγέ, Αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το αν κάποιο είναι πρόθυμος να αποκτήσει δεξιότητες κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σταδιοδρομίας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δούμε τι γίνεται στον τομέα των υπηρεσιών, στις μεταφορές, στις κατασκευέ. και αυτό που πρέπει να αλλάξει ε, στο εκπαιδευτικό μα σύστημα και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Θα υπάρχουν ε, επαγγέλματα, αλλά τι είδους επαγγέλματα είναι τα συστήματά μας αρκετά ευέλικτα. Ως πολιτικοί είμαστε έτοιμοι για δράση. Ελπίζω ε, όλοι σας να έχετε κάποιο χρόνο να μπείτε στη δική μας την ιστοσελίδα και να δείτε την, ε, τις αλλαγές που έγιναν το 2018 ε, αλλαγές ε, οι οποίες ε, δείχνουν ότι έχουμε ελπιδοφόρα τεχνική και περίπου 200 νέα επαγγέλματα. Είναι μια έκθεση που μας ανοίγει τα μάτια και δείχνει ότι αν είμαστε αρκετά επίσης με το εκπαιδευτικό μας σύστημα νομίζω ότι θα κερδίσουμε περισσότερα από τις αλλαγές που θα επέλθουν. Και ο συνήθως η ε, τεχνολογία είναι πολύ πιο γρήγορη από τις μελέτες, ε, κατά κανόνα και πολύ πιο γρήγορη από εμάς τους ε, πολιτικούς. Όταν μια μελέτη είναι έτοιμη, ήδη κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Κάθε χρόνο αλλάζει η τεχνολογία, η νέα έρευνα καθίσταται ήδη απαρχαιωμένη, άρα δηλαδή οι πολιτικοί μας ε, καλούνται να έχουν το θάρρος να στρέψουν το βλέμμα στο μέλλον και να αναζητήσουν λύσεις ε, οι οποίες ε, επιτρέπουν στο να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα για να καλυφθούν οι ανάγκες του κόσμου και κυρίως ε, της δουλειάς. Όταν εμφανίζεται κάτι καινούργιο, κατά κανόνα το πιο, σημαντικό, το πιο δύσκολο είναι να αλλάξει κανείς τη σκέψη. Και ως πολιτικός πρέπει να σας πω ότι για μας αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα πάντα κάνουμε πράγματα, ε, σκέπτονται οι άνθρωποι, γιατί να πρέπει να τα αλλάξουμε. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αλλάξει, ε, τι είναι εκείνο που πρέπει να αλλάξει στη Φινλανδία χρειαζόμαστε περισσότερους ε, ε, περισσότερα μαθήματα που να προσαρμόζονται σε ανθρώπους με έλλειψη δεξιοτήτων αλλά και ανθρώπων που ζουν μέσα στην ε, τεχνολογική επανάσταση. Περισσότερους κύκλους μαθημάτων για άντρες, για γυναίκες, για εργαζόμενους που χρειάζονται νέα προσόντα. Ε, πρέπει να αλλάξουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να στηρίξουμε την εκπαίδευση με έναν ευφυή τρόπο. Και κατ' ουσίαν χρηματοδοτούμε κάτι καινούριο το οποίο οδηγεί σε καλά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας. Ε, δεν είναι το να έχουμε μια τυχαία εκπαίδευση χωρίς να βλέπουμε τι πραγματικά χρειάζεται και ποιες είναι οι ανάγκες ε, της βιομηχανίας. Οφείλουμε να φτιάξουμε ισχυρούς μηχανισμούς ε, για να αποκτηθούν νέες δεξιότητες. Οφείλουμε να καταστήσουμε γνωστό το τι πρέπει να αλλάξει. Ε, οι συμβουλές για την ε, σταδιοδρομία του μέλλοντος. Αυτό σίγουρα το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μία μονοαπευθυντική θηρίδα αν θέλετε και ένα ε, πιο εύκολο σύστημα για την εκπαίδευση να μπορεί κανείς να εκπαιδευτεί διαδικτυακά ε, μέσα από πύλες και ιστοσελίδες ε, να μπορεί να εκπαιδευτεί με μεγαλύτερη ταχύτητα μελέτες για καλύτερη διαχείριση. Αυτά τα χρειαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα και επίσης και οι ηγέτες πρέπει να είναι έτοιμοι για το μέλλον. Χρειαζόμαστε και μεγαλύτερες περιόδους για την χάραξη πολιτικής, ε, αναλύσεις ε, ε, που να αφορούν ΜΚΟ, εταιρείε. Επίσης, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και για την ανάπτυξη των νέων κυρίως να ενισχύσουμε την κατάργηση των αποκλεισμών στις κοινωνίες μας. Η κυβέρνηση πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει ε, την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση έτσι ώστε να ενταχθούν περισσότερα περιθωριοποιημένα παιδιά. Και έτσι θα έχουν περισσότερα παιδιά πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάτι που ήταν πάρα πολύ δαπανηρό για πολλές οικογένειες ε, δωρεάν σχολικά βιβλία και πολλά άλλα. Και έτσι θα καταστεί δυνατόν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανισότητες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κατάλληλη στιγμή ε, ή σωστό να σταματήσω τώρα την παρέμβασή μου. Ας έχουμε μια επικοδομητική συνεδρίαση, μια ζωντανή ε, συζήτηση και να μάθει η μία από την άλλη πλευρά. Γιατί να κάνουμε συνεχώς και πάντα τα ίδια λάθη. Νομίζω ότι θα πρέπει πάντα να βρούμε τις καλύτερες ε, ιστορίες επιτυχίας ε, και κάποιες από αυτές να τις εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας. Το μέλλον πράγματι είναι μπροστά μας, αλλά εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ακόμα πολλά πράγματα και θα επιβιώσουμε των αλλαγών εάν μπορέσουμε να κοιτάμε προς το μέλλον και να ε, δραστηριοποιούμεθα με σοφία στην Ευρώπη αλλά και σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ακυλώνεν. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Άντε Μπάμπιτς από το Κρατικό Κοινοβούλιο είναι μέλος ε, της Επιτροπής Εργασίας Συνταξιοδοτικού Συστήματος και Κοινωνικής χιώσης Έχετε το λόγο κύριε Μπάμπιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μάρας. Αξιότιμη κυρία Χαραντσόβα, Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσω στα ακροατικά, στη μητρική μου γλώσσα. Είναι τιμή και προνόμιο να σας απευθύνω το λόγο σήμερα και να πω δύο λόγια για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ποιες δεξιότητες και ποιες θέσεις εργασίας απαιτούνται προκειμένου να δώσουμε μια όθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας ε, στο σημερινό κόσμο, ο οποίος είναι γεμάτος προκλήσεις. Η δυναμική τεχνολογική ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές αλλαγές και η γυράσκουσα κοινωνία έχουν αντίκτυπο σε πολλέ κοινωνικέ πτυχέ και φυσικά στον κόσμο τη εργασία. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε νέε τεχνολογίε, νέε τάσει, ε, ε, διαδικτυακά ζητήματα, τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ, ε, εικονική πραγματικότητα. Όλα αυτά έχουν αλλάξει τον τρόπο στον οποίο ζούμε και συνεργαζόμαστε. Το περιβάλλον εργασία και οι κοινωνικέ μα σχέσει υπόκεινται σημαντικέ αλλαγέ και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Στην Ευρώπη και στην Κροατία, η διαδικασία αυτή μεταφράζεται σε όλο ένα και μεγαλύτερη ανάγκη ε, εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς. Πέραν λοιπόν της τυπικής εκπαίδευσης, ο σύγχρονος ε, κόσμος της εργασίας αναζητά επιπλέον δεξιότητες και γενικές γνώσεις, αλλά και ψηφιακές δεξιότητες ε, και συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη, όπως επεσήμανε και ο κύριος Σμιτ. Μόνο ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό μπορεί να δώσει στην βιωσιμότητα και στην ανάπτυξη. Γι' αυτό ακριβώς ε, πιστεύω ότι πρέπει να ε, γίνει απαραίτητο επενδύσει σε ε, εκπαίδευση υψηλή ποιότητα. Θα πρέπει επίση να υπάρχουν πολιτικές της αγοράς εργασίας και διαβίου μάθηση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στι παρούσε προκλήσει. Το πρώτο βήμα είναι να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να περιλαμβάνει και επαγγέλματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασία. Καθώ καθώς επίσης και επαγγέλματα τα οποία θα αυξηθούν περισσότερο στο μέλλον, όπω ανέφερε και η Φιλανδή συνάδελφο. Υπ' αυτή την έννοια, η εταιρική σύμπραξη μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματο και τη αγορά εργασία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκια, πολλό δε μάλλον ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ε, κοινωνικών λειτουργών και των ε, εργοδοτών που πρέπει να ε, κάτσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι για να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πολιτικές απασχόλησης. Πρέπει επίσης να υπάρχει προσαρμογή και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρέχεται διαβίω εκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή στις αλλαγές αυτές, διότι η συνεγής εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού συμβάλλει στην μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και στην καλύτερη απασχολησιμότητα. Στη Δημοκρατία της Κροατίας ε, το σύστημα της διαβίου μάθησης είναι μάλλον κατακαιρματισμένο. Υπάρχουν ε, αλληλοεπικαλύψεις στι δραστηριότητε και αυτό που διαπιστώσαμε στο σύστημα είναι ότι δεν υπήρχε κατάλληλο συντονισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων και του εκπαιδευτικού συστήματο και τη απασχόληση. Γι' αυτό ακριβώ και συστήθηκε ένα φόρουμ για διαβίου επαγγελματική ε, καθοδήγηση και προσανατολισμό. Ε, συμμετέχουν υπουργεία, δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμοί, κοινωνικοί εταίροι, επιμελητήρια, ενώσει, συνδικάτα και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ε, πανε, πανεπιστημιακή κοινότητα και συνδεδεμένα επαγγέλματα. Ο στόχο είναι να προωθήσουμε το διαβίω επαγγελματικό προσανατολισμό ώστε να προέρχεται και διαβίω εκπαίδευση και κατάλληλε κοινωνικέ πολιτικέ. Χαίρομαι λοιπόν που το φόρουμ μα επισημαίνεται ω παράδειγμα καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέραν των αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα, στη διαβίω εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε και περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να έχουμε βιώσιμες ε, εργα... θέσεις οι οποίε θα είναι και και επίση να επενδύσουμε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και για τους νεότερους αλλά και για τους ε, μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους και όσοι βρίσκονται σε θέσεις απασχόλησης που αντιμετωπίζουν ε, αλλαγές στον οικονομικό τομέα εργασίας τους λόγω των ε, ταχύτητα των αλλαγών στην κοινωνία. Λόγω των δημογραφικών δικτών και της γύρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στους μεγαλύτερους ηλικία εργαζομένους που πρέπει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Επίσης πρέπει να παρασχεθούν και εκεί κίνητρα στους εργοδότες ώστε να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στις εργασίες και να είναι και μέντορες για τη νεότερη γενιά εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο η Κροατία τροποποίησε το νόμο για την ε, συνταξιοδοτική ασφάλιση ώστε οι συνταξιούχοι να μπορούν να εργαστούν και μετά την ηλικία συνταξιοδότησης αν το επιθυμούν. Στην Κροατία ε, σήμερα επιτρέπεται τετραήμερη εργασία σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων. Ε, τετράωρη, συγγνώμη, εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και επίση πρέπει να τονίσουμε ότι ε, είναι κοινή ευθύνη όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία, δημόσιου φορεί, εργοδότε, αλλά και του ίδιου του εργαζόμενου, καθώ επίση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω ανέφερε και ο κύριο Σμιτ. Θα πρέπει επίση να τονίσω ότι ο βασικό ρόλο του δημόσιου τομέα στην ανάπτυξη και προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματο και στην ανάπτυξη προγραμμάτων που είναι προσαρμοσμένες στις ε, ανάγκες της οικονομίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα και οικονομικά αλλά και μη Γι' αυτό ακριβώ και η Κροατική Προεδρία καλωσορίζει τι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικαιροποίηση του θεματολογίου για τι δεξιότητε για την Ευρώπη για την ενίσχυση τη εγγύηση για την νεολαία. Είναι επίση υπέρ τη εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που θα βοηθήσουν εργαζόμενου από κάθε γενιά να διαχειριστούν οι ίδιοι τη σταδιοδρομία του. Θα ήθελα επίση να τονίσω ότι η Κροατία είναι ένα από τα νεότερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής και έχει υποφοληθεί από ευρωπαϊκέ, ε, ε, πρωτοβουλίες για παράδειγμα παράδειγμα, η εγγύηση για την νεολαία. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντα ότι εγώ είμαι πεπισμένο ότι σε αυτό το πλαίσιο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν τι προσπάθειέ του στο σχεδιασμό εργαλείων που θα μα επιτρέψει να προβλέψουμε τι μελλοντικέ ανάγκε των εργαζομένων, καθώ επίση και ε, αποτελεσματικά εργαλεία για την. Ε, ε, αξιολόγηση των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο και στις ανάγκες, να υπάρχει κατάλληλη στήριξη, ευκαιρίες για κατάρτιση και εκπαίδευση, για να βελτιώσουν τις δυνατότητες τους είτε να βρουν μια καλύτερη θέση εργασίας ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, και εμείς ε, σας ευχαριστούμε. Η επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Κλάουδια Μίλα από το Γερμανικό Κοινοβούλιο ε, ε, μέλο τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργεια. Κυρία Μίλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να λάβω το λόγο, αλλά για να μην χαθώ και εγώ στη μετάφραση θα μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα, στα γερμανικά. Κυρίες και κύριοι, Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία ε, αρχική παρατήρηση. Όταν ήρθε η επανένωση, αυτό ήταν στα νέα κράτη, στα νέα κρατήρια μια πολύ μεγάλη αλλαγή και είχε επιπτώσεις όχι μόνο στην ε, κοινωνία αλλά και στα επαγγέλματα γιατί πάρα πολλά επαγγέλματα απλά ήταν άγνωστα και πολλά δεν χρειαζόντουσαν καθόλου. Ξαφνικά λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν μπροστά στο να πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα, να εκπαιδευτούν περαιτέρω και αυτό το άλμα στην εποχή δεν το κατάφεραν όλοι. Οι αλλαγές που βρίσκονται τώρα μπροστά μας ε, είναι γνωστές, ε, δεν είναι απρόσμενες, είναι τα θέματα της ψηφιοποίησης, ε, της κλιματικής κρίση. Ε, και όπως ελέγχθη χθε και πολύ ωραία η δημογραφική αλλαγή. Αυτές τις αλλαγές τις βλέπουμε και για το λόγο αυτό ε, μπορούμε να προσαρμόσουμε την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση μας. Στη Γερμανία εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές στο πώς ακριβώ ε, εννοεί κανείς την περαιτέρω κατάρτιση. Τα περισσότερα τέτοιου μέτρα λαμβάνονται στις επιχειρήσει, δηλαδή γίνονται, προσφέρονται από τους εργοδότες και πληρώνονται από τους εργοδότες. Και εδώ υπάρχουν ε, πολλές διαφορές ε, από ότι για τις ε, μικρές επιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πολλές ανάγκες αλλά πολλές φορές δεν είναι σε θέση να πληρώσουν και να αποδεσμεύσουν και τους εργαζόμενους. Επίσης και το, επίπεδο των, το τυπικό επίπεδο των σπουδών και αυτό παίζει ρόλο για τη περαιτέρω εκπαίδευση. Το 98% των ανθρώπων που έχουν σπουδάσει συνεχίζουν ε, όσοι έχουν μια απλή εκπαίδευση είναι το 46% και εκείνοι χωρίς δεξιότητες μόνο 34%. Άρα δηλαδή ακριβώς εκείνη η ομάδα στην οποία θέλουμε να απευθυνθούμε αυτή τη στιγμή με τα μέτρα μας δεν το καταφέρνουμε. Και επιτρέψτε μου και άλλη μία σύντομη παρατήρηση. Στη Γερμανία η εκπαίδευση δεν είναι εθνικό καθήκον, είναι καθήκον των κρατηδίων. Έχουμε λοιπόν ένα κατακαιρματισμένο σύστημα με διαφορετική πρόσβαση, διαφορετικό κόστος. Επιπλέον ε, πολλές φορές η παιδεία δεν είναι δωρεάν. Έχουμε ένα σύστημα όπου ε, μπορεί κανείς να συνδυάσει τη σχολική εκπαίδευση με την εκπαίδευση ε, στις επιχειρήσεις. Είναι το περίφημο διοικό σύστημα. Και εδώ συμβαίνει πολύ συχνά το εξής. Ε, η ε, αποζημίωση μετά από μετακπαίδευση δεν είναι τόσο εντυπωσιακή. Άρα δηλαδή το θέμα είναι πώς μπορούμε να προσφέρουμε κίνητρα έτσι ώστε όλοι να εκπαιδεύονται και να μπορούν μετά και να μετακπαιδεύονται. Στο Bundestag πρόσφατα βιώσαμε ε, και αποφασίσαμε μία αλλαγή ε, του συστήματος ενίσχυσης και στήριξης των φοιτητών. Υπάρχει αυτό το σύστημα στη Γερμανία, στηρίζονται οικονομικά όσοι θέλουν να μετεκπαιδευτούν. Βεβαίως, ε, πολλοί θα ήθελαν να προσφέρονται περισσότερα, κυρίως ε, εκείνοι που κάνουν μετεκπαίδευση να έχουν ουσιαστική οικονομική αποζημίωση και με τα χρήματα που κερδίζουν να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, να είναι κάτι το περιζήτητο η μετεκπαίδευση και να μην φοβάται κανείς ε, την ε, κοινωνική υποβάθμιση. Πολύ σωστά αναφέρθηκαν τα περίφημα One Stop Shop, μία ιδέα την οποία και εμείς τη συζητάμε για εκείνους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουν δουλειά. Το αντίστοιχο ε, γραφείο του ΑΕΔ, ας το πούμε έτσι, ε, αυτό είναι αρμόδιο για εκείνους όμως ε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν καθόλου απασχόληση. Τίθεται λοιπόν το εξή ερώτημα. Μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, να προσφέρουμε ευκαιρίες σε ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι. Μέχρι τώρα περισσότερο στίγμα αποτελούσε το να απευθυνθεί κανείς σε γραφείο του ΑΕΔ και να δηλώνει ότι χρειάζεται εκπαίδευση. Ε, κάτι άλλο επιπρόσθετο, το να μπορεί κανείς ε, να αποδεσμεύεται από την εργασία του, αυτό ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Παράλληλα όμως ο εργοδότης πρέπει να έχει και αυτός κάποιο όφελος, δηλαδή η μετεκπαίδευση να ωφελεί και τον εργοδότη. Και εφόσον συζητάμε για αυτά τα θέματα, ε, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και για τα επαγγελματικά παιδεία. Δηλαδή αυτά τα οποία διδάσκονται, αυτά τα οποία προσφέρονται ως μετεκπαίδευση είναι ακόμα επίκαιρα. Γιατί υπάρχει το θέμα της δημιουργίας νέων επαγγελμάτων τίθεται το ερώτημα κατά πόσον ε, παλαιότερα επαγγέλματα δεν έχουν εξαφανιστεί. Η συνάδελφος από τη Φινλανδία έθιξε το θέμα της κατάργησης των αποκλεισμών και αυτό έχει σχέση με την μετεκπαίδευση. Να ανοίξουμε το βλέμμα μακριά από τους ε, κλασικούς εργοδότες προς τους ανθρώπους ε, με ειδικέ δεξιότητες αυτοί να συμπεριληφθούν περισσότερο στο σύστημα και ε, αυτό εγώ το λέω πάντα να έχουμε κυρίως ε, στραμμένο το βλέμμα στις γυναίκες σε πάρα πολλούς ε, τομείς και επαγγέλματα αυτό δεν το κάνουμε επαρκώς πρέπει λοιπόν και εδώ να καταστήσουμε σαφές ότι ε, όσο δεν αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την ομάδα δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε και το πρόβλημα. Σήμερα το πρωί ε, τέθη το εξής ε, θέμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να συμπεριλάβουμε όλους τους πολίτες ε, στις αλλαγέ που γίνονται. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλους μας θα υπάρχουν προβλήματα. Οι άνθρωποι θα μας τρέψουν την πλάτη αν δεν έχουν τις ευκαιρίε ενός νέου ψηφιακού κόσμου. Η μετεκπαίδευση είναι ακριβώ το κλειδί για να φέρουμε με τη μεριά μα όλου αυτού του ανθρώπου. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μίλλερ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο σκέλος της συνεδρίασης, ανταλλαγή απόψεως μεταξύ των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο στην ε, Αντιπρόεδρο την κυρία Χαραντσόβα για να ε, συντονίσει αυτή τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαράς. Ε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του πάνελ για τα εισαγωγικά του σχόλια. Είμαι βέβαιη ότι ε, θα υπάρξουν αρκετές αντιδράσεις. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση να σας πω κάποια διαδικαστικά. Όπως γνωρίζετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπλε κάρτα σας αν θέλετε να λάβετε το λόγο. Ε, θα φροντίσω να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στη συζήτηση, αλλά θα ήθελα απλώ να σας υπενθυμίσω ότι η παρέμβασή σας θα πρέπει να είναι το πολύ τρία λεπτά. Και με αυτό να δώσω το λόγο στον κύριο Πέτρη από τη Γερμανία. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να σας πω ότι εγώ ε, προέρχομαι από μια περιοχή της Γερμανίας που θα την γνωρίζει ο κύριος Σμιτ. Είναι το Ζάρλαντ το οποίο εκλήθη να ε, αλλάξει πολλές αλλαγές ε, στο Ζάρλαντ σε τελική ανάλυση αυτό ε, κρίνεται ως κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά και σε εμά όπως και η κυρία Μίλλερ, τα στοιχεία δεν είναι πολύ καλύτερα. Πράγματι υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά τα δύο φύλλα. Και αυτό το βλέπει κανείς και στο τέλος της εργασιακής ζωής, όταν το ε, θέμα που τίθεται είναι η σύνταξη. Και βλέπουμε ότι η φτώχεια έχει θηλυκό πρόσωπο. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα, η διαβίου μάθηση είναι ένα από τα βασικά μέτρα ο εργασιακός κόσμος αναφέρθηκε αυτό, αλλάζει και εάν έχετε κανείς από μια περιοχή με άνθρακα και χάλιβα, ε, η κατάργηση των ανθρακοριχείων, η κρίση στην ε, χαλιβουργία, όλα αυτά ε, σημαίνουν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να είναι υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό λοιπόν κατά τη δική μου την άποψη είναι απολύτως απαραίτητο οι εργοδότες να ενδιαφέρονται κυρίως ε, για το ότι οι εργαζόμενοι τους ε, χρειάζονται μία προσφορά ε, επαγγελματικής κατάρτισης. Στη Γερμανία αυτό είναι και αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αυτό είναι και δικαίωμα του εργαζόμενου. Στη Γερμανία έχει κατατεθεί και μία πρόταση από το δικό μου κόμμα, από τους σοσιαλδημοκράτες, ε, γενικά αυτό να είναι ε, κατοχυρωμένο δικαίωμα. Όσο διαρκεί η εκπαίδευση, τρία χρόνια, αυτό σημαίνει είναι 12 ημέρες ε, στο σύνολο της εργασιακής ζωής. Αυτά για τη μετακπαίδευση. Άρα δηλαδή οι εργοδότες ε, θα πρέπει να εκπληρώσουν το κοινωνικό τους ε, καθήκον και να στηρίξουν τους εργαζόμενους. Επίσης είναι καθήκον του κράτους να δημιουργήσει το απαραίτητο πλαίσιο και τα πρότυπα που θα επιτρέπουν στον εργοδότη ε, να είναι αποτελεσματικό σε αυτά που προσφέρει και να προσφέρει ε, μετακπαίδευση και εκπαίδευση και στα δύο φύλλα. Εγώ θα ήθελα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν μέσα σε ένα ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτά να μην είναι μόνο ε, μια εθνική επιλογή αλλά να γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας δώσει ε, προτάσεις για ένα ελάχιστο πλαίσιο που πρέπει να υφίσταται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πέτρη και επόμενος είναι ο κύριος Στάροβιτς από τη Σλοβενία. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και θα μιλήσω σλοβενικά. Μία γλώσσα την οποία μιλούν δύο εκατομμύρια άνθρωποι. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω όλου σα. Θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι χαίρομαι ιδιαίτερω ότι μία από τι προτεραιότητε τη Νέα Επιτροπή είναι να δοθεί μεγαλύτερη επικέντρωση στο χάρτη των ανθρωπίνων κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει πιο πολύ αλληλεγγύη, πιο δίκαιη η Ευρώπη και πιο πολύ συνοχή. Χαίρομαι επίσης που θα υπάρχει πιο πολύ κοινωνική διάσταση στο οικονομικό μας σύστημα. Γιατί αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη ανάπτυξη και πιο βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη. Χρειάζονται, λοιπόν νέα προσέγγιση για την οικονομικές προκλήσεις. Ένα θέμα που έχει επισημάνει και ο ΣΑ και υπάρχει πιο πολύ επιστημονική βάση για την καλύτερη και βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη. Νέες τεχνολογίες λοιπόν και νέος ορισμός, νέοι ορισμοί σε ό,τι αφορά βιώσιμες πολιτικές, δημιουργικές πολιτικές. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν του ΩΣΑ διασυνδέεται με μια ευθύ στρατηγική και ένα παρτιτήριο και μια πολιτική για την ε, συμπεριληπτική ανάπτυξη. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Σλοβενία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αυτή και ε, είναι συμπρόεδρος μάλιστα σε μια ομάδα φίλων του προγράμματος. Η Σλοβενία έχει ακόμα οικονομική ανάπτυξη, αλλά δεν έχουμε επαρκές εργατικό δυναμικό. Δεν έχουμε τους εργαζόμενους εκείνους με τις απαραίτητες δεξιότητες. Έχουμε ένα κενό λοιπόν στην αγορά εργασία. Και αυτό γιατί, γιατί πάντα κοιτάμε το σκέλο τη αγορά και θεωρούσαμε ότι η αγορά θα ήταν η καλή λύση για όλα τα προβλήματα. Αυτό όμω είναι μια λύση η οποία είναι καταναγκαστική. Ο Πρωθυπουργό δήλωσε ότι δεν ανταποκρίνεται στις νέες αυτές προσεγγίσεις Ελπίζω ότι οι νέες επενδύσεις και στην επιστημονική ανάπτυξη θα μετατραπούν σε επενδύσεις στην κοινωνία για το πώς η κοινωνία και τα θεσμικά όργανα θα βρουν σωστές λύσεις για πιο πολύ αποτελεσματικότητα για να είναι πιο αποτελεσματική η κοινωνική Ευρώπη και η Ευρώπη στο συνολό Πολλά παιδιά σήμερα, αφού ολοκληρώσουν τη σχολική τους εκπαίδευση, θα εργάζονται σε ένα κλάδο ο οποίος ακόμα δεν υφίσταται. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον κύριο Σάροβιτς, επόμενος ομιλητής. Η κυρία Κρέτσο, από τη Ρουμανία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αγαπητοί φίλοι. Και είναι πολύ σημαντικό να διδαχθούμε οι μεν από τους δε και από τις εμπειρίες που έχει ο καθένας. Πολύ φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή που ζούμε και έχουμε εμπειρίες τις οποίες δεν είχε κανείς άλλο στο παρελθόν. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση περνάει από τον επιχειρηματικό κλάδο και αυτό θα γίνει ε, είτε συμφωνούμε είτε όχι. Δεν ε, τον νοιάζει πολύ τον επιχειρηματικό κλάδο σε ό,τι αφορά την πλήρη απασχόληση, τα θέματα κοινωνική ασφάλιση, τα συστήματα συνταξιοδότηση το θέμα των πόρων του προπολογισμού και του, της ιδιωτικής σφαίρας. Δεν είναι δική του αρμοδιότητα, δεν είναι δικό του καθήκον, αν θέλετε. Δικό μας καθήκον είναι. Η Ένωση δεν έχει ψηφιακή κυριαρχία. Αυτοί που μπορούν να ελέγχουν το σερβερ μας ελέγχουν πραγματικά το σκεφτόμαστε. Το είδαμε αυτό και στις ε, εκλογικές εκστρατείες και στα δημοψηφίσματα και στις εκλογές. Οι υπολογιστέ και η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσουν σταδιακά όλο και πιο πολλέ εργασίε που τώρα έκαναν οι άνθρωποι. Βασιζόμασταν στην ε, η προϋπόθεση ότι όλοι είχαμε μία θέση απασχόληση, πλήρη απασχόληση για μία ζωή, ότι είχαμε σύνορα για να περιορίσουν το κεφάλαιο, αλλά η ψηφιακή πραγματικότητα είναι εντελώ διαφορετική. Χρειαζόμαστε νέα κοινοτόμα μέτρα. Χρειαζόμαστε και παγκοσμίου κανόνε για τη νέα πραγματικότητα όπου δεν υπάρχουν σύνορα και φυσικά εξουσία για να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τη φορολογία, πολιτική βούληση επίσης. Αυτή η πολιτική βούληση ακόμα δεν υπάρχει και η σχετική ικανότητα για την εφαρμογή όλων αυτών, η οποία επίσης ακόμη λείπει. Να έχουμε επίσης υπόψη ότι ο έλεγχος δεν είναι πάντα αποτελεσματικό μέτρο, αλλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με θέματα εκπαίδευση, όπως είπαν πολλοί. Όχι μόνο για τα παιδιά, όχι μόνο για τους νέους. Διαβίου μάθηση για να αντιστέκεται κανείς για να προσαρμόζονται, να αλλάζει δουλειά, να σταματά, να αρχίζει, συγγνώμη, ε, ανεξάρτητες διαδικασίες αυτοαπασχολούμενων. Τα μέτρα όμως αυτά προϋποθέτουν να αλλάξουν οι προτεραιότητές μας σε ό,τι αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Και αυτό σήμερα, όχι σε 10-20 χρόνια, εδώ και τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μακάρα από την Κροατία έχει στη συνέχεια το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να γίνει ανταγωνιστική σε αυτή την ψηφιακή επανάσταση. Και καθώς αναπτύσσονται οι ψηφιακές ε, δεξιότητες ε, ε, θα ανοίξουν και οι θύρες της ψηφιακής οικονομίας. Η ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη δεν μπορεί να αναπτυχθεί εάν δεν αντιμετωπίσουμε το γεγονό ότι έχουμε σπάνιδα ψηφιακών δεξιοτήτων και αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε επανειλημμένο σήμερα. Οι ψηφιακέ δεξιότητε θα δημιουργήσουν νέε θέσει εργασία για όλου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων ήδη αποτελεί περιορισμό για την ανάπτυξη στην Ευρώπη οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν θέσει εργασία που του αξίζουν. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στι επιχειρήσει μα να έχουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ψηφιακών ταλέντων. Δεν υπάρχουν αρκετοί πολίτε στην Ευρώπη που να έχουν τι απαραίτητε ψηφιακέ δεξιότητε. Γι' αυτό και ακριβώ υπάρχουν θέσει εργασία οι οποίε παραμένουν κενέ σε πολλού τομεί. Ε, το ποσοστό τη ανεργία των νέων ανθρώπων μεταξύ 15 και 24 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 20%. Το 1 τρίτο του εργατικού δυναμικού έχουν μόνο τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το 45% του συνολικού πληθυσμού μάλιστα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε περίπου 1 εκατομμύριο νέους ανθρώπους προκειμένου να πληρώσουν θέσει εργασία στον ψηφιακό τομέα και αυτό θα πρέπει να γίνει με μαθητεία, πρακτική άσκηση, κατάρτιση και με βραχυπρόθεσμα προγράμματα απασχόλησης. Θα πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε τους εργαζομένους μας και θα πρέπει να τους επαναπροσανατολίσουμε και να επενδύσουμε στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε για τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων, για τη συμμετοχή στην αγορά εργασία και στην κοινωνία εν γέννη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι θέσει ε, πληροφορική και επικοινωνία παρέχουν πολλέ ευκαιρίε και σε άνδρες και σε γυναίκε και έχει ήδη ε, τονιστεί ότι υπάρχει ένα κενό και χάσμα μεταξύ των μισθών ανδρών και γυναικών και το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις. Υπάρχουν επίσης και ευέλικτα ωράρια εργασίας που είναι ε, είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός ε, για την ε, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Η καινοτομία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες επίσης θα μας δείξει και πόσο σημαντικό είναι να μάθει κάποιος νέες δεξιότητες γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σε νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και στον επιχειρηματικό κόσμο και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κούτρα Κουκουμά από την Κύπρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Των εργαζομένων στην Κύπρο είναι ανησυχητική και αντανακλά τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ που επιβάλλονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μερική απασχόληση έχει αυξηθεί σημαντικά σε βάρο τη μόνιμη απασχόληση, η αγορά εργασία έχει απορριθμιστεί, μεγάλων ποσοστών των εργαζομένων δεν καλύπτεται από συλλογικέ συμβάσει, οι νέοι της κύπρου οδηγούνται στη μετανάστευση προς αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης στο εξωτερικό το κράτος πρόνοιας έχει αποδομηθεί και συρρυκνωθεί. οι συντάξεις έχουν μειωθεί και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παραμένουν απροστάτευτες. Ο πίνακα κοινωνικών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων καταγράφει τι ιδιαίτερε προκλήσει στον τομέα τη απασχόληση, το υψηλό ποσοστό ατόμων που διαβιούν στο όριο ή κάτω από το όριο τη φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού καθώ και των ατόμων που βρίσκονται εκτό εκπαίδευση απασχόληση και κατάρτιση. το εισόδημα των νοικοκυριών είναι χαμηλότερο από το 2008 και το ποσοστό των εργαζομένων φτωχών είναι ανησυχητικό εδώ ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού και να εκφράσω την ανησυχία μου για το ενδεχόμενο να καταστεί ο δούριο ύπο για την ανατροπή των συλλογικών συμβάσεων και τη οργάνωση των εργαζομένων. εξάλλου το σύμφωνο για το ευρώ καθορίζει ως κριτήριο για τη διαμόρφωση των μισθών τη σχέση τους και με την ανταγωνιστικότητα. οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε και να απαντήσουμε το ερώτημα τελικά θα νοιαστούμε και θα επικρατήσει ο στόχος της ανταγωνιστικότητας ή το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων σε σχέση με τον κατώτατο μισθό αδύρυτη ανάγκη είναι επίσης η θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τις νέες μορφές ε, απασχόλησης προκειμένου οι εργοδότες να υποχρεώνται να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις την υλοποίηση ελάχιστων όρων απασχόλησης για τους εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις καθώς και μέτρα που να ενισχύουν την εργασιακή ασφάλεια η ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και εποπτείας είναι εκ των ουκάνευ για τη δημιουργία νέων ποιοτικών αξιοπρεπών θέσεων εργασίας με πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Εδώ θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου από όσα έχω ακούσει και από τον Επίτροπο αλλά και άλλους ομιλητές στο πάνελ όπως είναι ότι δεν θα υπάρχουν δουλειές για μια ζωή, ότι κάποιος θα μπορεί να αλλάξει επάγγελμα δέκα φορές στον εργασιακό του βίο ε, η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση που σίγουρα παραπέμπει στην επέκταση των ορίων συνταξιοδότησης και βέβαια το συνεχώς επαναλαμβανόμενο τη διαβίου εκπαίδευση που παραπέμπει ξανά στην εργασιακή ανασφάλεια στην ε, ελληνική ε, ιστορία υπήρχε πάντα η διαβίου εκπαίδευση που εσήμενε ή το γυράσκω αή διδασκόμενος που εσήμενε ότι ε, για όλη μου τη ζωή μορφώνομαι για να γίνω καλύτερος. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι δυστυχώς για να αλλάσω επάγγελμα που επιβεβαιώνει τη δυσχερή θέση που βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Thank you very much. The next speaker on my... Ευχαριστώ. Επόμενος, ε, ο κύριος Τούσεκ από την Κροατία. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν αναφερόμαστε στα σημαντικά αυτά θέματα και τις προκλήσεις αυτές που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά εργασία, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονό ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση. Γιατί κάθε νέα γενιά ε, χάνει σε πληθυσμό κατά 25% από την προηγούμενη. Οι, νέες, ε, οι νέοι θέλουν να φτιάξουν οικογένεια και να, και να συμμετέχουν στην ε, επαγγελματικό βίο, αλλά είναι δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, σε πολλά κράτη υπάρχουν προβλήματα με την φύλαξη των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανεί και να δουλεύει και να φροντίζει το παιδί του. Ένα άλλο θέμα είναι η έλλειψη χώρου στου βρεφονιδιακού σταθμού, ιδιαίτερα τα απογεύματα, η έλλειψη ευελεξία. για να προσαρμοστούν και οι εργοδότες στις ανάγκες των γονιών που εργάζονται. Και αυτό προφανώς ε, συνήθως ε, αποβαίνει βάρος των γυναικών, γιατί αυτές είναι αυτές που θυσιάζονται αν δεν υπάρχει κάποια θεσμική μορφή φύλαξης. Δεν είναι προς το συμφέρον τους, προφανώς, ε, των εργοβατών να δώσουν ε, πλεονεκτήματα και προτίμηση στις νέες γυναίκες με παιδιά, εάν δεν αναγκαστούν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντικές είναι οι πολιτικές ε, υπέρ της γεννητικότητας για να υπάρξει υποστήριξη του συστήματος. Χρειάζεται λοιπόν να αναλάβουμε ε, τις ευθύνες μας στον τομέα αυτό για να δημιουργήσουμε όρους που θα είναι φιλικοί προς τις οικογένειες. Επίσης και ευρωπαϊκά ταμεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κίνητρα για τις εταιρείε προκειμένου να εισαγάγουν αυτά τα φιλικά προς τις ε, οικογένειες μέτρα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Σίκουτ από την Εστονία για το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμφίβολα ε, οι δεξιότητες, η μετεκπαίδευση, ευκαιρίες μετεκπαίδευσης, η ελεύθερη πρόσβαση, τα μαθήματα online, τα προσαρμοσμένα μαθήματα, αυτά είναι απολύτως απαραίτητα και όλα συμβάλλουν στην μετάβαση που χρειαζόμαστε μια μετάβαση που θα μας φτάσει στο ψηφιακό και πράσινο μέλλον. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι είναι απαραίτητο να δουλέψουμε και στο μυαλό των ανθρώπων, όπως είπε και ο Επίτροπος Σμιτ. Βλέπουμε ότι η μετεκπαίδευση δεν είναι υποχρέωση, είναι μια ευκαιρία. Ευκαιρία για τους ανθρώπους ε, όσον αφορά τη δουλειά και το εισόδημα, αλλά ε, επειδή οι άνθρωποι με υψηλότερη εκπαίδευση είναι πολύ πιο πιθανό να συμμετέχουν στη διαβίου μάθηση, οφείλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα εμπόδια και τα κίνητρα σχετικά με τη διαπίου μάθηση. Παραδείγματο χάρη, ε, το Ταμείο Ασφάλισης ε, στην, ε, στην Εστονία συμπεριλαμβάνει και όσους έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο και τι αποκτούν νέες δεξιότητες μέσα από τη δουλειά, ε, μαθαίνουν ε, από τους γονείς τους, όμως ε, δεν θεωρούν τους αυτούς τους φοιτητές. Και όλες οι εκστρατείες οι οποίες γίνονται, οι μελέτες, η συμμετοχή στη διαβίου μάθηση, αυτοί που συμμετέχουν ε, δεν έχουν κατά νου τις εκστρατείες γιατί ε, δεν θεωρούν ότι είναι ο στόχος αυτών των προγραμμάτων. Έχουν αρνητική εμπειρία στο σχολείο, στην ε, μάθηση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση έτσι ώστε όσοι χρειάζονται τη μετεκπαίδευση να την αποκτήσουν, να μπορούν και αυτοί να κατανοήσουν ότι παρότι παρελθούσα εμπειρία τους μπορεί να είναι αρνητική, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή ότι τα προγράμματα δεν τους αφορούν. Γι' αυτό λοιπόν ας ε, ασχοληθούμε με την προσέγγιση των ανθρώπων και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε ένα πιο ευφυές και πιο ψηφιακό εργατικό δυναμικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Περές από την Ισπανία, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω ισπανικά. Έχω δύο παιδιά, 8 και 12 ετών και είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι όταν θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας δεν θα είναι ε, με μια δουλειά η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αν κάνουν ένα παραδοσιακό επάγγελμα, αν επιλέξουν ε, είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν γιατί θα εργαστούν κατά πάσα πιθανότητα σε κάτι που δεν υπάρχει. Όταν ετέθη σήμερα ε, το θέμα, ε, το σωστό ερώτημα είναι πώς βλέπουμε ε, τον εκπαιδευτικό κόσμο σε ένα τέτοιο δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. Δόθηκαν αρκετές απαντήσεις και κάποιες τις είδα με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα κίνητρα για να συμμετέχει κάποιος στην αγορά εργασία με πίστοση στην κατανάλωση, όπω γίνεται στη Γερμανία. Πρέπει οι νέοι όχι μόνο να έχουν μια θεωρητική κατάρτιση που θα του επιτρέπει ε, να έχουν κάποιε δεξιότητε, αλλά όσο εκπαιδεύονται σε θεωρητικό επίπεδο, να μπορούν να συμμετέχουν και στον πραγματικό κόσμο ε, τη εργασία και να μαθαίνουν κάτι καινούριο. Αυτό δεν είναι καινούριο. Το λέμε στην περιοχή τη Εστρεμαδούρα από το 2014 και λειτουργεί με αποτέλεσμα. Ε, είμαι από την Ισπανία που είμαστε ηγέτε στην ανεργία στην Ευρώπη και μάλιστα στην ανεργία των νέων. Τα στατιστικά στοιχεία όμως λένε ότι έχουμε την γενιά των νέων με την καλύτερη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Επομένως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτού που αναζητούν οι εργοδότες και αυτού που σπουδάζουν οι φοιτητέ και μπορούν να προσφέρουν. Μπορεί να είναι πιο μορφωμένοι λοιπόν οι νέοι μα, αλλά δεν έχουν αυτό που αναζητούν οι επιχειρήσει. Τεχνητή νοημοσύνη, blockchain και όλα τα συναφή, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει φτάσει. Θα πρέπει να τα αναπτύξουμε όλα αυτά με ευρύ τρόπο. Η πρόκληση στην Ισπανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμω είναι να μπορέσουμε να κάνουμε αυτέ τι συνδέσει. Να δώσουμε στου νέου στην Ευρώπη ικανότητε που θα τους κάνει ελκυστικού για εργοδότε σε όλο τον κόσμο και να είναι πολύ σημαντικέ και οι γλώσσε στην κατάρτισή του τα παιδιά μα, όπω είπα στην αρχή, θα εργαστούν σε θέσει εργασία που ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό σημαίνει ότι για να το επιτύχουν αυτό πρέπει να εκπαιδεύσουμε του νέου μα στι νέε τεχνολογίε και να του βοηθήσουμε να εργαστούν στην αγορά εργασία και να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία που μόνο η εργασία σου δίνει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει ήδη από τώρα. Το τελευταίο έτος του ορίζοντα 2020 πρέπει να είναι αυτό το ε, συνδετικό στοιχείο για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τους νέους μας για τις δουλειές του μέλλοντας. Ας εργαστούμε λοιπόν από εδώ ώστε το Είναι υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη από χώρα σε χώρα. εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει πιο πολύ αποτελεσματικότητα, η οποία θα σημαίνει να αυξηθούν οι μισθοί και όχι να υπάρχει ε, εξίσωση προς τα κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να συνεχίσουμε άλλο έναν ε, βουλευτή από την Ισπανία, τον κύριο Σάντσο, στα Ισπανικά, η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και θα μιλήσω Ισπανικά. Καλησπέρα σε όλους σας. Η πολιτική μου ομάδα, Vox, το κόμμα μου, είναι μάλλον στην ε, ομάδα του ECR των ε, μεταρρυθμιστών και στερετικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρούμε ότι το θέμα της εκπαίδευσης έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου και γι' αυτό λοιπόν οι δημόσιες ε, αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα δημόσια θεσμικά όργανα και τα ιδιωτικά, ιδιωτικέ οργανώσει θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση για του νέου, προκειμένου να αναπτύξουν μέσα στον τρόπο την ε, τεδρομία του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή εκπαίδευση και των ατόμων ε, στη δευτεροπάθμια εκπαίδευση, γιατί σε κάποιες χώρες όπως στην Γαλλία για παράδειγμα ξεκινάμε μια κοινή βάση και στη συνέχεια καλύπτονται πολλά στοιχεία. Και όλοι οι μαθητές στις χώρες αυτές λοιπόν θα πρέπει να καλύπτουν τέσσερις τομείς. Ο πρώτο τομέας έχει να κάνει με την ε, εκμάθηση της εθνικής γλώσσας. Αυτό είναι θέμα πολιτισμού. Το, θέμα, το δεύτερο, ο είναι οι φυσικη και οι φυσικές επιστήμες, ιδιαίτερα στα μαθηματικά, προκειμένου να μπορέσει ο κάθε μαθητής να σκέφτεται και αφηρημένα και να μπορεί να κατανοήσει τις φυσικές συνδέσεις που υπάρχουν. Κατά τρίτον, προσφέρεται μία επιπλέον γλώσσα πέρα από τη μητρική, μία ξένη γλώσσα δηλαδή, προκειμένου να μπορεί κανείς να κατανοήσει και τις κουλτούρες άλλων κρατών και τέλος μία βασική εκπαίδευση ε, στα ψηφιακά ζητήματα. Αυτά τα τέσσερα λοιπόν στοιχεία είναι εκ των ΟΚΑΝΕΦ. για να αντιμετωπίσουμε την ε, έλλειψη εκπαίδευση η οποία μπορεί να προκύψει από την ε, ψηφιακή υπερεξειδικευσή. Εγώ είμαι πανεπιστημιακό καθηγητή εδώ και 30 χρόνια και τα διαπιστώνω όλα αυτά. Έχω προσωπική εμπειρία. Αλλά τίθεται θέμα ε, γενική παιδεία, το οποίο θα πρέπει ουσιαστικά να ισχύει για όλου. Δεν τίθεται θέμα μόνο οικονομικής αξιοποίησης. Τίθεται θέμα ανθρώπινη αξιοπρέπειας. Και αυτό συνάδει απόλυτα με μια εξέλιξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε ό,τι αφορά την οικονομική πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε. Αυτές λοιπόν οι δεξιότητες θα πρέπει να προωθηθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα πρέπει αυτό αυτό όλα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της δυτικής οικονομίας. Γιατί η δυτική οικονομία είναι αυτή η οποία δημιουργεί τις πιο πολλές θέσεις απασχόλησης. Αυτές λοιπόν οι δεξιότητες θα πρέπει να αναπτυχθούν και επί της βάσης αυτής θα πρέπει να βελτιωθεί και η επαγγελματική κατάρτιση. Δεν πρέπει να υπάρχουν ανισότητες όπως παρατηρούνται σε πολλές χώρες όπως για παράδειγμα στην Ισπανία. όπου έχουμε πολλά πανεπιστημιακά διπλώματα, αλλά αυτά τα πτυχία δεν χρειάζονται απαραίτητα στην οικονομία. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια τεράστια απογοήτευση για του φοιτητέ, γιατί όταν αποφοιτούν δεν έχουν πού να απασχοληθούν. Για την ανθρώπινη λοιπόν ε, αξιοπρέπεια δεν χρειάζεται πανεπιστημιακό δίπλωμα. Χρειάζεται μία αξιοπρεπή δουλειά, ένα αξιοπρεπή μισθό και να εκτιμά η κοινωνία την εργασία που εκτελεί το άτομο ανεξάρτητα από το αν συνοδεύεται με πτυχίο ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και Και έτσι ολοκληρώνεται ο κατάλογο των ομιλητών. Και στο σημείο αυτό θα δώσω το λόγο πάλι στους πανελίστες. Νομίζω ότι ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα σχόλια και πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από διάφορα τμήματα της Ευρώπης και μέρη της Ευρώπης. Νομίζω ότι ένα θέμα ήταν κοινό ο αντίκτυπο τη ε, ψηφιακή ε, επανάσταση στην αγορά εργασία. Και μια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δημοσίευσε σήμερα τι πρώτε ανακοινώσει για τα ψηφιακά, θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχά στον εκπρόσωπο της Επιτροπής και να μας ε, κάνει και κάποια σχόλια καταλεκτικά. Έχετε το λόγο κύριε Επιτροπέ. Ο κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Και έχετε το δίκιο. Η μεγάλη πρόκληση είναι η ψηφιακή πρόκληση. Γιατί αυτή η πρόκληση θα αλλάξει κατά πάσα πιθανότητα το μεγαλύτερο τμήμα των θέσεων απασχόλησης. Και αυτό θα σημαίνει ότι όλοι μας θα πρέπει να επενδύσουμε στις γνώσεις αυτές. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν το οποίο θα ήθελα να επαναλάβω είναι το εξή. Η επένδυση στη γνώση, η επένδυση στη διαβίου μάθηση, αυτά αποτελούν θετικά στοιχεία. Δεν είναι μια υποχρέωση, ένας περιορισμό, είναι μια νέα ευκαιρία. Θα πρέπει λοιπόν να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα σε όλου όσοι ανησυχούν, ανησυχούν δικαίω για το ποιο θα είναι ο αντίκτυπος της ψηφιακή αυτής επανάστασης τη της απασχόλησης. Αυτό που έχουμε να τονίσουμε όμως είναι ότι δεν είναι μόνοι του αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει όλοι οι υπεύθυνοι στο δημόσιο τομέα, τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και αυτή, αλλά και ο ιδιωτικός κλάδος, όλοι λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουν το πλαίσιο της διαβίωματισης. Η ψηφιακή ανάπτυξη, επανάσταση λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε και την προπτική μας αλλά και την διάστασή μας. και κάτι το οποίο αποτελεί πραγματικά πρόβλημα και το οποίο συγκρατώ είναι ότι αυτοί οι οποίοι είναι οι λιγότερο καλά εκπαιδευμένοι είναι εκείνοι στους οποίους επενδύουμε λίγο, λιγότερο. Και παρόλα αυτά, οι δικέ του θέσει απασχολήσεις είναι αυτές που απειλούνται πιο πολύ από κάθε άλλε. Άρα το διακύβευμα είναι να βρούμε, κάποιο το ανέφερε άλλωστε, να βρούμε τις καλύτερες μεθόδους προκειμένου αυτοί οι εργαζόμενοι, αυτοί οι υπάλληλοι, αυτοί οι εργάτες να στραφούν προς την κατάρτιση και όντως πολλοί εξ αυτών δεν έχουν ε, πολύ θετική εντύπωση από το σχολείο. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν νέους τρόπους για την εκπαίδευση, την κατάρταση, για να δώσουμε νέες προπτικές στους ανθρώπους αυτούς και νέες ευκαιρίες. Και αυτό αποτελεί μια επανάσταση κατά κάποιο τρόπο, γιατί θα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο της εκπαίδευσης. Τρίτο σκέλος. Συχνά είναι οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι εκείνοι. Όταν μιλάμε για ηλικιωμένου, μιλάμε συχνά για νέους ανθρώπους ακόμα. Σε αυτούς λοιπόν είναι πιο, γίνονται πιο λίγες επενδύσεις. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ε, μια ψηφιακή διάσταση. Ρίξει στι εταιρείε προκειμένου να, υπάρξει, να υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση στα άτομα αυτά. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε τέτοια διακριτική μεταχείριση. Όταν μιλάμε για διαβιμάθηση, θα πρέπει να μιλάμε πραγματικά για όλη τη ζωή του κάθε εργαζόμενου. Α, μη σας πω και μετά τη λήξη της επαγγελματική του σταθερομίας, γιατί αυτή η ιδέα της ε, ενεργούς γύρανσης ε, που προωθείται είναι σημαντική. Θα πρέπει και μετά τη σταδιοδρομία του κανείς να έχει πρόσβαση στη διαβίωμα Σήμερα λοιπόν διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες όντως έχουν μικρότερη παρουσία στις νέες τεχνολογίες. Περίεργο όμως, γιατί όταν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα ε, των κοριτσιών και των αγοριών στο σχολείο, τα κορίτσια διαπρέπουν πιο πολύ σε σχέση με τα αγόρια μεταξύ άλλων και στα ψηφιακά. Και παρόλα αυτά, όταν έρχεται η στιγμή να βρουν ε, μια θέση απασχόληση, μια δουλειά, υπάρχει ζήτημα. Το θέμα λοιπόν της ισότητας των φύλων έχει να κάνει και με την ψηφιακή αυτή μετάβαση, με την ψηφιακή αυτή αλλαγή. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το εξή. Τα επόμενα χρόνια, και όταν λέω τα επόμενα χρόνια δεν εννοώ σε 20-30 χρόνια, μιλάω τα επόμενα 5, 7, άντε 10 χρόνια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε, να επανεκπαιδεύσουμε παραπάνω από το ίμιση e των ε, εργαζομένων. Μιλάμε για 100, 120, 130 εκατομμύρια ανθρώπους. Μιλάμε για ένα τεράστιο διακύβευμα και ένα σημαντικό διακύβευμα και από οικονομικής άποψης. Όπως αναφέρθηκε, δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς δημόσια χρηματοδότηση, χωρίς επενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Και μιλώ για επενδύσεις. Επένδυση στην ε, δεξιότητα, στη γνώση. Είναι εξίσου σημαντική αυτή η επένδυση, όπως και η επένδυση σε μηχανήματα, σε ρομπότ. Θα πρέπει να αλλάξουμε επίσης και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοιες επενδύσεις στο εσωτερικό των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες εκπαίδευσης. Και προφανώς και σε επίπεδο δημοσιονομικής ε, πολιτικής και προλογίας. Σε κάποιες εβδομάδες θα έχουμε λοιπόν αυτή τη νέα ατζέντα για τις ε, δεξιότητες. Πρόκειται για ένα ε, πρώτο βήμα. Και προφανώς αυτή η ατζέντα θα πρέπει να μεταφραστεί ανάλογα με τις εμπειρίες, την κουλτούρα της ε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε χώρα, είτε είναι πιο γρήγορη, είτε είναι πιο αργή σε κάποια ζητήματα. Και σύμφωνα με τι ιδιαίτερε απαιτήσει που θα προκύψουν, για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, θα μεταμορφώσει το περιβάλλον στι ε, επιχειρήσει, τον ε, τρόπο παραγωγή. Θέματα όπως η υγεία, όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να προετοιμαστούμε για τις αλλαγές αυτές. Αλλά πάντα με αυτοπεποίθηση. Όχι να προκαλούμε φόβο στον κόσμο. Θα πρέπει να του δώσουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Γιατί θα αλλάξουν δουλειά για καλύτερες θέσεις απασχόλησης, με λιγότερο βαθμό δυσκολία, σε λιγότερη ε, χαρακτήρα επανάληψης. Γιατί αυτό στο οποίο διαπρέπουν οι άνθρωποι είναι η δημιουργικότητα, η συνεργασία και στο επίπεδο αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι παίζουμε το μέλλον μας σε επίπεδο επιχειρήσεων. Έχουμε μια σημαντική στρατηγική για το ψηφιακό κόσμο και από την επιτυχία της στρατηγικής αυτής θα εξαρτηθεί το πώς θα τοποθετηθεί η Ευρώπη στο διεθνές προσκήνιο σε ό,τι αφορά το διεθνή και παγκόσμιο ανταγωνισμό ε, εναντί των ανταγωνιστών μας, ε, τον ΗΠΑ, της Κίνας, και των άλλων ανταγωνιστών μας. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στον άνθρωπο, στους άνδρες και στις γυναίκες, στα παιδιά. Χτες έγινε μία συζήτηση για την εγγύηση για τα παιδιά. Όλα αυτά στέκουν. Είμαι αισιοδόξο. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να την κερδίσουμε τη μάχη αυτή για να μεταμορφώσουμε την Ευρώπη, η οποία σήμερα αποτελεί μεγάλη οικονομική δύναμη και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει έτσι και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για το θετικό σας μήνυμα και τα ενταρρυντικά σας λόγια και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Κιλόνεν. Ε, στην εισαγωγή σας είπατε ήδη ότι πρέπει να μάθει μία από την άλλη πλευρά ε, και νομίζω ότι είχαμε αρκετές παρεμβάσεις από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να ε, μας πείτε κι εσείς τι ακριβώς συμπεράνατε από τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχω μάθει κάτι και είναι πολύ σημαντικό για τους πολιτικούς αυτά που έχω μάθει. Οι δικές μου οι παρατηρήσεις σχετικά με την ψηφιακή εποχή, εγώ όταν τις σκέφτομαι, σκέφτομαι ποιος κάνει τις αλλαγές. Μερικές φορές ε, έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι ε, δεν είναι πια κομμάτι όλου αυτού ότι όλα αυτά μοιάζουν σαν να έρχονται από το διάστημα κάπου μακριά από ένα μυστήριο χώρο και ε, κατ' ουσίαν όμως ε, εμείς ε, επιφέρουμε τις αλλαγές εμείς ε, είμαστε εκείνοι που λαμβάνουμε τις αποφάσεις, εμείς είμαστε εκείνοι που αποφασίζουμε αν θέλουμε η σκληρή δουλειά να είναι πιο εύκολη ή αν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Τελικά όμως ε, ε, ποια είναι η κατάσταση. Πώς ε, αντιμετωπίζουμε την ψηφιακή εποχή και όλα αυτά είναι καλά ή κακά. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγχει κανείς ψηφιακά θέματα από ότι την κλιματική αλλαγή. Μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας, ε, αλλά ε, όσον αφορά την φύση και τον πλανήτη, πάντα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από το να ελέγξει κανείς την ψηφιοποίηση ή να προσφέρει στους ανθρώπους ε, νέες ικανότητες. Εύχομαι και ελπίζω να αλλάξουν και τα πρότυπα ε, της κατανάλωσης. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν περισσότερες εμπειρίες, ε, κάτι διαφορετικό για τη ζωή τους, και νομίζω ότι αυτό είναι επίσης και μία ευκαιρία για τον τομέα παροχής υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν όταν οι άνθρωποι σκέπτονται ότι δεν υπάρχουν πια δουλειές για αυτούς νομίζω ότι ο τομέας της παροχής υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια θα κάνει άλμα, ίσως βέβαια να μην το έχουμε ακόμα αυτό συνειδητοποιήσει, γιατί εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα περισσότερα αγαθά μας καθιστούν καλύτερους ανθρώπους και ίσως την επόμενη χρονιά ή τα επόμενα χρόνια να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε διαφορετικά. Δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά τα καταναλωτικά προϊόντα. Δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε περισσότερο. Χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό που θα αντικαταστήσει την κατανάλωση στη ζωή μας. Και σήμερα ακούσαμε πολλές σημαντικές ε, ομιλίες για το τι τις ευκαιρίες υπάρχουν για να αποκτήσει κανείς ε, μάθηση. Τώρα το να προσπαθήσει κανείς να εκπαιδεύσει ανθρώπους ε, ε, χωρίς να τους ρωτήσει τι χρειάζεστε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στους ανθρώπους και να έχουμε ε, μαθήματα πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ανθρώπων. Και στην Ευρώπη το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ε, έχουμε γυράσκοντα ε, πληθυσμό και έλλειψη μωρών όπως ε, είπε και ο συνάδελφος πολύ σωστά έχουμε ξεχάσει την οικογενειακή ζωή εξακολουθούμε να θέλουμε οικογένειες να έχουμε ένα ευέλικτο σύστημα και να κάνουμε και ορισμένα άλλα πράγματα όχι μόνο να δουλεύουμε και θα ήθελα να τελειώσω τις παρατηρήσεις μου λέγοντας ότι ε, πρέπει να προσφέρουμε ελπίδα ε, στους απογοητευμένους, δεξιότητες ε, στους μη εκπαιδευμένους και να εμφυσίσουμε εμπιστοσύνη αντί για δυσπιστία. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε όλοι μας. Νομίζω η συζήτηση είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ταξιδέψουμε από το βορρά στο νότο. Είχαμε αρκετές παρεμβάσεις από την Νότια Ευρώπη, είχαμε αρκετές παρεμβάσεις από την Κροατία. Επομένως φαίνεται ότι το θέμα αυτό είναι υψηλά στις προτεραιότητες στην Κροατία. Είναι πολύ σημαντικό για την Προεδρία που είναι θετικό και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπάμπιτς για να δούμε αν συμφωνεί και με τις απόψεις της Φιλανδής συναδέλφου. Έχετε το λόγο. Κυρία Χαραντσοβά, φυσικά και συμμερίζομαι αυτές τις απόψεις και τα είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, αλλά ήταν πολύ καλό που ακούσαμε και τις παρεμβάσεις πολλών συναδέλφων που μίλησαν για το δυναμικό χαρακτήρα της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Όταν λέτε ότι καταγόμαστε από την Νότια Ευρώπη, όπου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού προς χώρες ε, όπου το βιωτικό επίπεδο είναι υψηλότερο και υπάρχουν ε, ε, περισσότερες θέσεις εργασίας, ο κύριο Στάροβιτ από τη Σλοβενία είπε ότι σήμερα η αγορά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά μας και το 65% αυτών που αποφυτούν από τα πανεπιστήμια λαμβάνουν ε, πανεπιστημιακούς τίτλους για θέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον. Από την άλλη ακούσαμε την κυρία Κουκουμά από την ε, Κύπρο που είπε ότι ο κατώτατος μισθός ε, θα πρέπει να ε, αυξηθεί και εξέφρασε τις ανησυχίες της και είπε ότι δεν θα μάθουμε και παλά όταν αρχίζουμε να ζητάμε από τους συνταξιούχους να συνεχίσουν να δουλεύουν. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν ακόμα το δικαίωμα να εργάζονται και μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασία και θα μπορούν ακόμα να αντικαταστήσουν το νεότερο εργατικό δυναμικό και να ε, είναι και μέντορες για αυτούς οι οποίοι ε, είναι νεοσερχόμενοι στην αγορά εργασία. Έχουμε τη διαβίω εκπαίδευση επίσης, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και το εξής. Ο κύριος Σμιτ στην εισαγωγή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αναφέρθηκε στην αναβάθμιση αλλά και στην νέα διαβάθμιση. Η αγορά εργασίας είναι δυναμική, δεν είναι στατική και ο κόσμος αλλάζει και ε, είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνεται μια νέα διαβάθμιση, να γίνεται αναβάθμιση, να υπάρχει διαβίου εκπαίδευση. Η κυρία Μίλουρ από τη Γερμανία είπε ότι κάποια πράγματα μπορεί να ισχύουν για κάποιες χώρες και κάποια άλλα όχι. Αυτό που είναι καλό σε αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να μας βοηθήσουν να λάβουμε κάποιες πληροφορίες. Και οι νέοι άνθρωποι μέσω της εγγύησης για την νεολαία η οποία θα δώσει το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες εργασίας και σε ίσους μισθούς. Αυτό είπε και η κυρία Φόντερ Λάιον στην ε, ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που έγινε αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι αυτά που είπε ο κύριος Σμιτ ε, στην αρχική του παρέμβαση Είναι κάτι μεν που συζητιέται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά θα πρέπει να συζητηθεί και στα εθνικά κοινοβούλια. Ό,τι συζητούμε εμεί στη χώρα μα θα συμβάλλει και στην οικονομία όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γεγονό ότι ω χώρα ε, γυράσκουμε ως πληθυσμός γενικότερα γυράσκει ο πληθυσμό και με τη βοήθεια ε, του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για τα δημογραφικά ζητήματα θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα ε, εργαλεία ώστε να έχουμε υψηλό ε, υψηλή ηλικία θνησιμότητας και να επιτύχουμε πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλύτερα σας σχόλια. Και τελευταίος, η κυρία Μελίρα από τη Γερμανία. Αν ρωτιέμαι, πού θα βρείτε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών που είπατε και των παρεμβάσεων που ακούσαμε ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παρόλο που έχει περάσει η ώρα. Η πρώτη μου εντύπωση είναι η εξή. Όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι η μετεκπαίδευση είναι πιο σημαντική παραποτέ. Είναι εκεί που θα κρυθεί, κατά πόσον η Ευρώπη θα ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του μέλλοντος, κατά πόσον θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε πραγματικά παντού την διαβίωμαθεση και την εκπαίδευση. Ακούσαμε διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία. Κατά πόσον είναι αυτό καθήκον καταρχάς του ιδιωτικού κλάδου ή του δημόσιου κλάδου για την εκπαίδευση, την επίσημη εκπαίδευση, έχουμε να πούμε το εξή. Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση στι πιο πολλέ ε, χώρε. Στον τομέα τη επαγγελματική κατάρτιση δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο. Θα ανακύψει λοιπόν το ερώτημα και θα έπρεπε να το εξετάσουμε το ερώτημα αυτό. Θα πρέπει να κινηθούμε προ την κατεύθυνση αυτή η μετακπαίδευση είναι ένα δικαίωμα για μια ολόκληρη ζωή και τι θα σήμαινε αυτό. Θα σήμαινε στην πράξη ότι θα έπρεπε να διαθέσουμε τις απαραίτητες υποδομές. Θα σημαίνει αυτό άραγε ότι ο επαγγελματικό ε, κόσμος και τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να προσαρμοστούν. Εδώ συμφωνώ με τον συναδελφό από την Κύπρο. Για πολλούς είναι ε, πολύ τρομακτικό το να αλλάζει ε, κανεί θέση απασχόληση, να αλλάξει διαρκώ ε, δουλειέ, αλλά αποτελεί και μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι κίνδυνο. αν ε, δεν έχω τη δυνατότητα να προσαρμοστώ στις αλλαγέ αυτές. Αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο καθήκον ε, της αγορά. θα πρέπει να είναι και καθήκον της, του κράτου. Γιατί το κράτος είναι αυτό που θα χάσει, η Ευρώπη είναι αυτή που θα χάσει αν δεν εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις ευκαιρίες αυτές και η συνάδελφος από την Εστονία δυστυχώς έφυγε. Είπε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε ακριβώς τα άτομα αυτά που δεν ε, συμμετέχουν στην διαδικασία μετεκπαίδευση και διαβίου γιατί αυτοί απειλούνται για τον ε, συνάδελφο από την Ισπανία για το θέμα της εκμάθησης γλωσσών στο σχολείο. Φυσικά πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα της εκμάθησης ε, δεξιοτήτων για τον υπολογιστή στα ψηφιακά. Αυτό που λείπει είναι η δημιουργικότητα, η δυνατότητα κριτικής ε, εξέτασης όλων των στοιχείων και αυτές είναι οι σημαντικές προτεραιότητες στην ε, καινούργιο ψηφιοποιημένο κόσμο. Η κυρία Μαρκάλ το είπε ξεκάθαρα το ερώτημα και το θέμα του κατά πόσον θα επικρατήσουν τα fake news, ή ε, ψεύδεις αυτές ειδήσει. είναι και θέμα εκπαίδευσης. Είμαστε σε θέση να αμφισβητήσουμε αυτά που πρέπει να αμφισβητήσουμε στον ψηφιακό κόσμο, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε σε επίπεδο κοινωνικό. Δεν είναι θέμα μόνο της οικονομίας, είναι θέμα κοινωνίας. Αυτό είναι το θέμα. Το κατά πόσον θα συνεχιστούν όλα αυτά και θα μπορέσουν να υλοποιηθούν σε μια καλή και δυνατή Ευρώπη ή κατά πόσον θα διασπαστούμε. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη. Γιατί έχουμε μια παρέμβαση της τελευταίας στιγμής. Θεσμικό ζήτημα. Η κατα ποσον θα διασπαστουμε ευχαριστω και ζητω συγγνωμη γιατι εχουμε μια παρεμβαση τη τελευταια στιγμη θεσμικο ζητημα η επιτροπη των Περιφερειών ζήτησε το λόγο από τον κύριο Κρατσιόνα εισηγητή για τι κοινωνικέ πολιτικέ. Ένα λεπτό. Ο κ. Καρατσόνα έχει το λόγο. Thank the... Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συμπρόεδροι των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων, Έρχομαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, από την ε, συνέλευση της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, εμείς αποδίδουμε σημασία στην βελτίωση του θεματολογίου για τις δεξιότητες με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης δεξιοτήτων και της δίκαιης μετάβασης. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό το θεματολόγιο είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Πρέπει να υπάρχει επικαιροποίηση με αναφορά στις τοπικές και τις περιφερειακές ε, προϋποθέσεις ε, και τους υπάρχοντες ε, πόρους. Το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο, είναι μια κοινωνική επένδυση. Ε, γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει αναβάθμιση των δεξιοτήτων ε, όταν δεν το ζητούν αυτό οι ίδιοι εργαζόμενοι. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία με βάση τις εταιρικέ σχέσεις ανάμεσα στις εθνικές, τις περιφερειακές αρχές, τις εταιρείε ε, και επίσης και τους παίκτες της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος είναι να αποκτηθούν περισσότερες δεξιότητες μέσα από άτυπα ε, και, ε, μη τυπική, και τυπική εκπαίδευση. Για να δώσω ένα παράδειγμα, από το τοπικό επίπεδο έχουμε ένα πρόγραμμα εμεί το οποίο εφαρμόζουν ε, οι δήμοι και οι κοινότητες στην Ουγγαρία. Για τους Ρωμά, πάνω από 100 Ρωμά απέκτησαν πλήρη απασχόληση στο δημόσιο τομέα με εργασίες από συντήρηση κτηρίων μέχρι την Κυπουρική. Το πρόγραμμα προσέφερε πολλές δυνατότητες ε, και αλλαγή προσέγγιση σε σχέση με την απασχόληση. Επίσης, ε, το πιστοποιητικό ε, έδωσε, προσέφερε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους εργαζόμενους και μάλιστα ανελήφθησαν και κάποιες πρωτοβουλίες για την βελτίωση των δεξιοτήτων κάποιων υποομάδων. Αυτά όλα κατέληξαν στο να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των οικογενειών. Ήταν λοιπόν μια εξέλιξη όπου όλοι κέρδισαν με ένα πρόγραμμα μικρής κλίμακας. Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο καθίσταται όλο και πιο σημαντικό στο να υπάρχει διαχείριση δεξιοτήτων. Πολλές φορές υπάρχει μια πιο ε, καινοτόμα προσέγγιση και θεσμική υποστήριξη. Δύο θέματα εδώ είναι πολύ σημαντικά. Η αφέμαξη εγκεφάλων και η ε, δημογραφική, αλλαγή. δημογραφική ε, αλλαγή. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι που απορρέουν από την διαρροή των εγκεφάλων. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή των Περιφερειών προτείνει ένα μηχανισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντονίζονται τα μέτρα για την διαρροή εγκεφάλων γιατί πρέπει να εξεταστούν όλες οι πτυχές εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εγώ είμαι συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις. Ε, αναβάθμιση λοιπόν των δεξιοτήτων. Αυτή είναι η βασική μας απάντηση στις προκλήσεις που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς ε, πάρα πολύ και νομίζω ότι τώρα πλέον ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας. Ε, θα ήθελα να ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή σας. Πριν λοιπόν ολοκληρώσουμε θα ήθελα εκ μέρους ε, όλων μας να ευχαριστώ τον συμπρόεδρό μου, τον κύριο Μάρας και θα ήθελα να του δώσω το λόγο για τις πραγματικά τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω εσάς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φιλοξενήσατε αυτή την κοινοβουλευτική εβδομάδα. Ήταν τιμή για μένα που συμμετείχα και που μπόρεσα να συμπροεδρεύσω. Ε, και εγώ θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα για να κάνω ανακεφαλαίωση κάποιων πραγμάτων, τα οποία κατά την άποψή μου είναι πολύ ε, σημαντικά. Τελειώνοντας αυτή η συνεδρίαση θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τις ε, παρεμβάσεις σας, κυρίως ε, όσους συμμετείχαν στο πάνελ που ήταν πάρα πολύ καλή για άλλη μια φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το θέμα αυτό ως ε, κάτι το οποίο πρέπει να βρίσκεται πολύ ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων της αμέσως επόμενης περίοδου. Ίσως να μην έχουν όλα τα κράτη-μέλη τις ίδιες προτεραιότητες όσον αφορά την κατάσταση στην παιδεία, ε, τις δεξιότητες ε, στην αγορά εργασίας. Αλλά σε τελική ανάλυση ε, όλοι ζούμε σε μία ένωση που διαμορφώνει από κοινού το μέλλον της. Επενδύουμε στους ανθρώπους, τα παιδιά, στο μέλλον και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να κατανοήσουμε ως προτεραιότητά μας. Πρέπει να πω από όλες τις συζητήσεις αν κατέληξα σε κάτι και μπορώ να το προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι όλες οι δράσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν ταχύτατα. Μόλις εντοπίσουμε κάτι, να αντιδράσουμε ταχύτατα. Παραδείγματο χάρη, όταν συνειδητοποιούμε ή πριν από κάποια χρόνια συνειδητοποίησαμε ότι υπήρχε πρόβλημα απασχόλησης, τότε η Επιτροπή πρότεινε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, το οποίο ήταν αποτελεσματικό στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τον ε, ίδιο δρόμο. Όταν μιλάμε για την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την αγορά εργασία βλέπουμε ότι δυστυχώς οι, πόλη μας, οι πολίτες μας στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις ε, δεν εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και αν δείτε λιγάκι ε, τους ε, απασχολούμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 10% αυτών έχουν μια επίσημη, ε, μια τέτοια εκπαίδευση που τους επιτρέπει να βελτιώσουν τη θέση τους. Βέβαια η κατάσταση σε ορισμένα κράτη είναι καλύτερη από άλλα, αλλά νομίζω ότι το 10% έτσι κι δεν αρκεί και κάτι άλλο που πρέπει να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι με χαμηλή εκπαίδευση κατά κανόνα οι άνθρωποι αυτοί δεν μπαίνουν σε μετεκπαίδευση. Μόνο ένας στους 25 με περιορισμένες δεξιότητες ε, χρησιμοποιεί ε, την διαβίου μάθηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της αυτά τα κρίσιμα θέματα που απαιτούν την ήπια εφαρμογή που και αυτή θα οδηγήσει σε καλές λύσεις. Και τέλος, δεξιότητες για όλους είναι κάτι που θεωρώ ότι είναι σημαντικό ε, για την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ε, κοινότητα η Ένωση που θέλουμε να έχουμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους ε, πολίτες μας να μπορούν και αυτοί να χρησιμοποιήσουν τη διαβίου μάθηση αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό ε, θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι θα υπάρξουν και πολλές άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε το θέμα αυτό στο μέλλον. Θα εξετάσουμε τις τάσεις, τις εξελίξεις και νομίζω θα μπορέσουμε να αλληλοβοηθηθούμε γιατί από κοινού μπορούμε να έχουμε ε, αγορά εργασίας υψηλότερου επίπεδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κράτη-μέλη θα επωφεληθούν, όλοι οι πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Well, this is it. <laughs> Αυτά λοιπόν είχαμε και σας εύχομαι καλό απόγευμα.